Το επόμενο θέμα στη μέση διάταξη αφορά το βασικό θέμα της χρηματοδότησης των μεταφορών του ψηφιακού τομέα, της ενέργειας και φυσικά την αναθεώρηση του μηχανισμού διασύνδεσης. Η έκθεση αυτή θα συζητηθεί και θα κριθεί ε, μέσω κοινών ε, συνεδριάσεων τραν ήτρε. Χαιρετίζω λοιπόν την παρουσία των συναδέλφων από την Ήτρε. Καλώς ήρθατε. Έχουμε λοιπόν χωριστεί μέρες διάταξη γι' αυτό. Αυτές οι κοινέ συνεδριάσεις θα προεδρεύονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ήτρε, ο οποίος δεν είναι παρόν αλλά ε, αναπληρούται. Και βεβαίως από μένα. Και Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Παουλ Ρούμπιχ που είναι εδώ για αυτή την συζήτηση και τον παρακαλώ, ε, αν το επιθυμεί, να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ την ε, πρόεδρο Ντελή. Εκπροσωπώ σήμερα τον ε, πρόεδρο Μπούζεκ Ξέρετε ότι η συνεργασία των δύο επιτροπών μας είναι θαυμάσια. Νομίζω ότι έχουμε ήδη αρκετή πείρα από αυτήν. Έχουμε πολλά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Οι δύο επιτροπές μας συνεργάζονται αποτελεσματικά και οι τρεις ε, εισηγητές τόνισαν ότι και για το θέμα αυτό έχει λειτουργήσει πολύ καλά συνεργασία Βίρκονεν, ε, ε, Μάριαν Μαρινέσκου και Πάβελ Τελίτσκα. Νομίζω ότι μέσω αυτής της συνεργασίας ε, αποδεικνύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει τους στόχους της. Αυτό είναι σημαντικό εν ώψη των ευρωεκλογών και ιδιαίτερα για το θέμα λοιπόν της ε, ενεργειακής απόδοσης που είναι στο κέντρο των προσπαθειών μας γιατί ιδιαίτερα ο τομέας των μεταφορών βλέπουμε ότι ε, Μπορεί να προωθηθεί λοιπόν η ενεργειακή απόδοση μέσω αυτής της ε, προσπάθειας για τη συνεχή ε, μετακίνηση, τη συνεχή κίνηση, να μην χρειάζεται να σταματάμε, να φρενάρουμε και να επιταχύνουμε συνέχεια. Ξέρουμε ότι έχουμε πολλά προβλήματα ε, λόγω του φρεναρίσματος έχουμε πολλά προβλήματα με τα πολύ μικρά σωματίδια διότι η τριβή που προκαλείται από το φρενάρισμα παράγει δισεκατομμύρια τέτοιων ε, ε, σωματιδίων. Βεβαίως για το ενεργειακό πακέτο η Ήτρε έχει επιτύχει πολλά και θέλουμε τη συνεργασία της ΕΣΑ, της ΕΝΙΖΑ και της ΜΠΕΡΕΚ. Η οριζόντια συνεργασία, συνεργασία και για τα δίκτυα TEN στον τομέα των μεταφορών θα βοηθήσει. Και βεβαίως Θέλουμε να υπάρξει πραγματική ψηφιακή εσωτερική αγορά. Τα 42 δισεκατομμύρια τα οποία αναφέρει το ε, CEF θα βοηθήσει η Ευρώπη να προωθήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της. Σε ευχαριστώ πολύ και να σας ξαναδώσω πάλι την Προεδρία, κυρία ε, Ντέλιε. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας. Χαιρετίζω την παρουσία και της ε, εισηγήτριας της Επιτροπής Περιφερειών. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Στο τέλος συζήτησης θα σας δώσω και ένα λεπτό για να μας πείτε τι ε, πιστεύουν οι περιφέρειες. Το πρώτο θέμα της κοινή μας ε, συνάντηση μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Και ξεκινάμε αμέσω με το θέμα αυτό που είναι ο μηχανισμός διασύνδεσης. Να ξεκινήσω τη συζήτηση και να δώσω το λόγο στον εισηγητή της Επιτροπής Τραν, τον κύριο, μάλλον του εισηγητέ ε, της Επιτροπής Τραν, Μαρινέσκου και Τελίτσκα και μετά την κυρία Βίρκουνεν από πλευρά Ήτρε για να μας υποβάλουν το σχέδιο έκθεση. Και κατόπιν θα έχουμε συζήτηση με τα μέλη που έχουν εγγραφεί. Κύριε Μαρινέσκο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Ρίμπιχ για την παρουσία του. Και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που έχουν συμβάλει στην εκπόνηση του σχεδίου έκθεσης. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία που ελπίζω να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες μέχρι να καταλήξουμε επί του θέματος αυτού. Έχετε δει τις προτάσεις μας. Θα αναφερθώ σε ορισμένα θέματα. Θέλω όμως να σας πω ότι δεν συζήτησα με τον κύριο Τέλιτσκα. Μέχρι στιγμή είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσω και μαζί του περαιτέρω. Αυτά λοιπόν που θα σας παρουσιάσω Ω, ναι, ναι, πολύ καλή συνεργασία μέχρι στιγμή, βεβαίω. Και νομίζω ότι θα συνεχιστεί. Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα υπάρχει. Είμαι βέβαιο. Λοιπόν, αυτά που θα σας πω λοιπόν μέχρι στιγμής είναι οι δικές μου απόψεις. Για τον προπολογισμό υπάρχει ένα προηγούμενο που εισήχθη από τους εισηγητές του πολιτούς πλαισίου για το Κοινοβούλιο για το πώς αντιμετωπίζονται όλες οι εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις για οριζόντια θέματα εν ώψη της ενδιάμεσης έκθεσης που θα υποβληθεί το Δεκέμβριο. Πολύ καλή διαδικασία, θεωρώ. Μας έδωσαν λοιπόν ορισμένες ενδείξεις. Ευχαριστώ τον κύριο Ρικέ για την γνωμοδότησή του. Ζητάει περισσότερη χρηματοδότηση αλλά παραμένουμε στο ίδιο ποσό για το υπάρχον CEF. Προτείνω να αυξηθεί το ποσό αυτό για να επανέλθει στο ποσό που πρότεινε το 2011 η Επιτροπή. 20 δις. Δηλαδή, εάν η Κομισιόν θεωρούσε πριν από 7 χρόνια ότι χρειαζόμαστε 20 δισεκατομμύρια για τις μεταφορές, τότε πρέπει να επαναφέρουμε αυτό το ποσό. Και είμεθα εντός του πλαισίου της διαδικασίας που προτείνουν οι εισηγητές Όλμπριχτ και Τομά για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όπως είπα λοιπόν το 2011 είχαν προταθεί 20 δις. Αλλά περιεκόπη πολύ λόγω της συζητήσεις με τον Κάμερο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τώρα έχουν αυξηθεί κάπως οι χρηματοδοτήσεις για τα ψηφιακά, επαρκώς για την ενέργεια, θεωρώ, αλλά για τις μεταφορές προτείνονται λιγότερα από το ισχύον ΣΕΦ. Αυτή είναι η πρότασή μου. Θα τη συζητήσω με τους συναδέλφους. Δεύτερον, η πρόταση για την πολιτική συνοχή είναι πολύ περίεργη. Αυτό το έχω ήδη συζητήσει με τον κύριο Τελίτσκα. Περίεργη λοιπόν πρόταση για την χρήση των ποσών που θα μεταφερθούν από την πολιτική συνοχή. 70% θα πάει για το ε, φάκελο που είναι για την πολιτική συνοχή και το 30% και το 30% συγγνώμη, θα πάει για το Rail Baltica. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε από ένα φτωχό κράτο μέλος για να δώσουμε σε ένα άλλο φτωχό κράτο μέλος. Γιατί ξέρετε ότι η πολιτική συνοχή, η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχή βασίζεται στο ΑΕΠ της κάθε περιφέρειας. Τα ποσά αυτά που είναι εντό του εθνικού ε, συνολικού πακέτου δεν μπορούν να μεταφερθούν ακόμη και εντό τη πολιτική συνοχή σε άλλο κράτο μέλο. Θα προτείνω λοιπόν την απάλληψη του σημείου αυτού από την έκθεση. Και το τρίτον, για το κράτο δικαίου. Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε όλες τι οριζόντιες εκθέσεις στο κράτος δικαίου. Υπάρχει ένας κανονισμό που εξετάζεται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο. Θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η αναφορά και στο ΣΕΦ, αλλά να τονίσουμε ότι αν πρέπει να ε, σεβαστούμε το κράτος δικαίου, θα πρέπει να σεβαστούμε και τις αναχώρα συστάσεις. Στο ίδιο επίπεδο να αναφερθούν δηλαδή αυτά τα δύο. Να εισαγάγουμε λοιπόν αυτό το στοιχείο στο σχέδιο εκθέσεις. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μαρινέσκου και ευχαριστούμε που τηρήσατε το χρονομιλία σας. Κύριε Τέλιτσκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, παρατήρησα την πρόκληση του κ. Βαντάλεν προς τον κ. Μαρινέσκου όσον αφορά τη συνεργασία ε, μέχρι στιγμή σας, σας ε, διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε την καλή μας συνεργασία. Υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των τριών μας και πάντα είναι ευχάριστο να συνεργάζεται κανείς με ανθρώπους που έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης. Τα καταφέρνουμε πολύ καλά, πιστεύω. Τι έχει γίνει τώρα μέχρι στιγμή, ε, το κείμενο που έχετε μπροστά σα, Υπάρχουν φυσικά κάποιε διαφορέ μεταξύ μα ε, που ακόμη δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Όπω ε, είπε και ο κύριο Μαρινέσκου, απομένουν 7 σημεία. Κατά βάση θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα πρώτο προσχέδιο ε, που σας προσφέρουμε ε, και μετά θα επιταχύνουμε με διάφορες τροπολογίες ε, για να απαλείψουμε τις κάποιες διαφορές που έχουμε και για να δούμε και κάποια σημεία όπου χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο. Περιλαμβανομένων των σημείων στο οποίο εστιάστηκε και ο Μαριάννα, τα οικονομικά τα κοιτάμε από διάφορες διαστάσεις, το συνολικό ποσό, την μεγαλύτερη απόδοση ε, και αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα και τη σύνδεση μεταξύ των τριών κυρίων τομέων. Δεν είναι μόνο θέμα συγχώνευσης, αλλά και καλύτερη χρήση όλων των κονδυλίων που υπάρχουν στη διάθεσή μας. Θα πρέπει να κάνουμε πολλά για να είμαστε αποτελεσματικοί και για το συνολικό ποσό πιστεύω ότι θα καταφέρουμε με τον Μαριάν και, και τη Χάνα να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Και βάσει των όσων είπε ο Μαριάν είναι σαφές. Ε, πρόκειται για μια επιτυχία μεγάλη. Το ΣΕΦ είναι επιτυχές, αλλά μπορεί να απλοστευτεί περαιτέρω, να φέρει και καλύτερα ακόμα αποτελέσματα βάσει των όσων βλέπετε μπροστά σα και άλλων προσπάθειων που θα κάνουμε. Χρειάζεται περισσότερη απλούστευση. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να παράσχουμε και κίνητρα στα κράτη-μέλη. Για πρώτη φορά θα παρατηρήσετε δεν επιβάλλουμε κυρώσει. αν υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση και επαφή μεταξύ των τομέων αν υπάρχουν διασυνοριακά έργα, κοινοπραξίες όπως τις ονομάζουμε που αποσκοπούν στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό, στην, οικοδόμηση, στην κατασκευή και στην υλοποίηση. Εκεί τα αποτελέσματα πιστεύουμε θα είναι καλύτερα και τα ωφέλη θα είναι μεγαλύτερα επίσης ε, μέσω της ε, συγχρηματοδότησης. Η Κομισιόν έχει εστιαστεί ιδιαίτερα στην συγχώνευση στο συνδυασμό πόρων, αλλά, αλλά δεν αρκεί ο πολιτικός λόγος. Πρέπει να γίνουν πράγματα στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να ε, είμαστε βέβαιοι ότι αυτός ο συνδυασμός, αυτό το blending είναι εφικτός, ε, ότι είναι αλληλοσυμπληρωματικός ε, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Τα περισσότερα έργα στα οποία αναφερόμαστε εδώ είναι έργα ειδικότερα στους σιδηροδρόμους που μας αρέσει ή όχι δεν είναι κερδοφόρα. Οπότε θα πρέπει να δούμε τα διάφορα οικονομικά μέσα που έχουμε, τα οικονομικά εργαλεία και πέραν της διευκόλυνσης συνδέοντας στην Ευρώπη, τι υπάρχει, τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό είναι άλλο ένα ζήτημα που εξετάζουμε. Στην πρόταση της Κομισιόν υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα διαιρέσει το Κοινοβούλιο και τις Επιτροπές, ε, το στρατιωτικό σκέλος, τα στρατιωτικά είδη, εγώ θα έλεγα είδη διπλής χρήσης. Είναι θέμα διπλής χρήσης εδώ. Αυτό δεν είναι ότι έχουμε ιδιαίτερη κατηγορία για τα στρατιωτικά προϊόντα. Ε, θέλω να σας διαβεβαιώσω, μιλάμε για μεταφορά και υποδομές ε, για μη στρατιωτικά Σκοπού σκοπούς για τα προϊόντα αυτά. Βάσει των όσων λέγονται ε, στα διάφορα έγγραφα και σε αυτή την ε, πρόταση με γνώμονα πάλι την καλύτερη αποτελεσματικότητα και την επιδεύξη των στόχων. Όπως είπε ο Μαριάν, απομένουν κάποια ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν μεταξύ των δυο μας, των τριών μας και υπογραμμίζω ότι ε, πράγματι έχουμε εξετάσει και οι τρεις σε διάφορες συναντήσεις αυτή την έκθεση συνεδριάζοντας μαζί. Πρέπει να το δούμε διασυνοριακά και διατομεακά. Είναι πολλά τα ζητήματα στα οποία θα πρέπει να σημειώσουμε κάποια πρόοδο μέσα στις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Θα επανέλθουμε με περισσότερες τροπολογίες, αλλά σίγουρα βλέπετε ότι εδώ υπάρχει μια ενοιολογική προσέγγιση, κάποιο όραμα, ε, όπως ελπίζουμε, επί χάρτου και αναμένουμε να ακούσουμε τα σχόλιά σας που θα μας βοηθήσουν να ρυθμίσουμε τις λεπτομέρειες ε, της πρότασης. Κάποιες από τις ιδέες που έχω δεν θα σας αναλύσω αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι πρώτα θα πρέπει να ενημερώσω τους συνεισηγητές μου, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουν και οι Διεπιτροπές με ένα άριστο αποτέλεσμα. Θα σας ευχαριστώ κύριε Τελετσικά. Ε, κυρία Βερικόνη τώρα έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Anymore how to use machines, you know. Ευχαριστώ, ναι. Βρήκα να ανοίξω και το μικρόφωνο μετά τι τελευταίε διακοπέ, δεν είναι αυτονόητο. Αγαπητοί πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω του συνεισηγητέ. Εγώ είμαι εισηγητρία από την Επιτροπή Γητρε. Ε, στο θέμα αυτό θα επικεντρωθώ στην ενέργεια και στον ψηφιακό τομέα, γιατί οι συνεισηγητέ μου μίλησαν ήδη για το σκέλο των μεταφορών. Και ο κύριος Τελίτσικα είπε ότι είναι εξαιρετική η συνεργασία. Ναι, όντω είναι κοινή η έκθεση και άρα και οι τρει θα πρέπει να βρισκόμαστε σε μια συμφωνία. Από πλευρά τη Επιτροπή ΙΤΡΕ, προφανώ οι μεταφορέ και η συνδεσιμότητα είναι σημαντικό σκέλο γιατί προαγάγει και την ανταγωνιστικότητά μα και τη βιομηχανία μα. Το... Η διευκόλυνση για τη συνέντευξη στην Ευρώπη παίζει σημαντικό ρόλο. Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικέ είναι οι επενδύσει αυτέ για την ενιαία αγορά και προκειμένου να υπάρχει ανταγωνιστικότητα και μια σύνδεση στην Ευρώπη. Η διευκόλυνση της Ένωτας στην Ευρώπη δίνει έναυσμα στις ε, υποδομές της ε, διευρωπαϊκές. Αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον. Και η τρέχουσα πρόταση λοιπόν ε, αυτή για το ΣΕΦ, όπως και προηγούμενη, έχει το τρεπλό αυτό σκέλος, Στην μεταφορές και την ενέργεια και τις υποδομές. Το νέο στοιχείο είναι η κινητικότητα στο στρατιωτικό τομέα και επίσης ένα νέο τομέα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ένα καινούριο στοιχείο στο πρόγραμμα αυτό. Επίσης έχουμε φιλοδοξούς στόχους για τους στόχους ε, για το κλίμα. 60% του, της χρηματοδότησης του ΣΕΦ έχει να κάνει με προγράμματα για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Πολύ φιλοδόξος ο στόχος, αλλά προφανώς είναι και πολύ σημαντικός ο στόχος που επιδιώκουμε. Στο πρόγραμμα λοιπόν ε, ΣΕΦ είναι σαφές τι προγράμματα μεταφορών χρηματοδοτούνται. Έχουμε τα TNT, έχουμε και στον τομέα της ενέργειας ε, τα δίκτυα TEN-E ενέργειας και έχουμε και τα project, τα προγράμματα κοινού συμφέροντος. Όπως θα θυμάστε, ψηφίστηκαν τέτοια προγράμματα ενεργειακά πρόσφατα. Έχουμε ένα κατάλογο λοιπόν των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα SEF Κοιτώντα δε και το πώ έχει λειτουργήσει τους τα τελευταία χρόνια, χρηματοδοτούμε μεγάλα προγράμματα για αγωγούς αερίου. Τα επόμενα χρόνια θεωρώ ότι θα έχουν τελειώσει τα μεγάλα αυτά προγράμματα, θα έχουν ολοκληρωθεί πλέον και άρα θα στραφούμε πιο πολύ στον ηλεκτρισμό και στη διασύνδεση ηλεκτρισμού. Αυτό προφανώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί διαρκώς αυξάνουμε τι ανανεώσιμε πηγές ενέργεια και εδώ χρειάζονται λοιπόν καλέ συνδέσει και διασυνδεσει για να υπάρχει και υποστήριξη του στόχου μεγάλων των διαδικτύων. Από πλευρά τη ενέργεια λοιπόν και από πλευρά των μεταφορών είναι σαφέ τι είδου προγράμματα χρηματοδοτούνται. Σε ό,τι αφορά το ψηφιακό σκέλος, έχουμε τα θέματα ανάπτυξης δικτύων 5G για την διασυνδεσιμότητα, ε, τη συνδεσιμότητα Gigabit και το ψηφιακό λοιπόν σκέλος ενδεχομένω να μην είναι τόσο συνεκτικό όσο τα άλλα δύο σκέλη. Ξέρουμε ότι όταν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη πλήρους συνδεσιμότητας, πρέπει να επενδύουμε σε πολλούς κλάδους ψηφιοποίησης. Άρα η αλλαγή που επιφέρει το τρέχον πρόγραμμα, το νέο μάλλον πρόγραμμα σε σχέση με το τρέχον, είναι ότι επικεντρωνόμαστε μόνο στην ψηφιακή υποδομή, στις ψηφιακές υποδομές. Τώρα έχουμε το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, όπου ε, χρηματοδοτούμε και άλλα ψηφιακά προγράμματα. Εδώ λοιπόν επικεντρωνόμαστε μόνο σε ψηφιακές υποδομές. Θέλαμε όμως να ξεκαθαρίσουμε τι είδου προγράμματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο ψηφιακό σκέλος. Γι' αυτό λοιπόν στην τροπολογία 30 κάνουμε μια πρόταση για να οριστούν τα προγράμματα κοινού συμφέροντος στο ψηφιακό σκέλος λίγο καλύτερα, γιατί πιστεύουμε ότι στο θέμα της ψηφιακής συντασιμότητα, αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι τα προγράμματα αυτά που συμβάλλουν ε, σημαντικά στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει και της Εθνικής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και που θα δώσουν και τις υποδομές που θα υποστηρίξουν τελικά τη μετάβαση αυτή προς την κοινωνία της διασυνδετισμότητας. ξέρουμε ότι αυτό το νέο πρόγραμμα θα συνεχίσει τη δουλειά που εγινε ο ρολος των συνεργειων γιατι ξερουμε οτι αυτο το νεο προγραμμα θα συνεχισει τη δουλεια που κανουμε στα πλαίσια του τρέχοντος προγράμματος, οτι θα χρηματοδοτήσουμε στην ενδιάμεση αναθεώρηση προέκυψε ότι θα έπρεπε να δείξουμε μεγαλύτερη βάρος ε, στις συνεργές. Γι' αυτό λοιπόν επικεντρωνόμαστε πιο πολύ στην εξέβρεση συνεργειών μεταξύ ε, μεταφορών ενέργειας και ψηφιακής ε, αγοράς. Αυτό προφανώς επηρεάζει και τους στόχους για την αλλαγή του κλίματος. Τα δίκτυα 5G στα μεγάλα δικτύα μεταφορών και οι εναλλακτικέ χρήσει εναλλακτικών καυσίμων αποτελούν πολύ καλά παραδείγματα του πώ συνενώνεται η ενέργεια, ο ψηφιακό κόσμο και μεταφορέ. Τέτοιου είδου προγράμματα θέλουμε για το μέλλον. Και εδώ θα επικεντρωθούμε λοιπόν πιο πολύ στο μέλλον. Όπως ξέρετε το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σφιχτό προθεσμία για κατάσταση τροπολογιών σε κάποιες εβδομάδες. Θέλουμε να ψηφίσουμε τον Οκτώβριο στην ε, κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών και αυτό πολύ φιλόδοξο στόχος, ε, αλλά ξέρουμε όλοι για ποιο λόγο γίνεται αυτή η υπερπροσπάθεια. Προσβλέπω στις συζητήσεις των δύο επιτροπών και προσβλέπω και στι τροπολογίε τι οποίε θα καταθέσετε εντό κάποιων εβδομάδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βρικούνα και θα ξεκινήσουμε λοιπόν πάρα αυτά τη συζήτηση με τους κοιόδους συζητητέ. και θα σα προειδοποιήσω ότι δύο λεπτά έχετε και μόνο αν δεν έχετε ολοκληρώσει πολύ απλά θα σα διακόπτω. Κυρία Αγιάλα Σέντερ, δύο λεπτά επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ πολύ τους συζητητές <clears throat> αυτή της πρώτης ε, εξέτασης Συμφωνώ με όσα υπόθηκαν. Να επανέλθουμε τουλάχιστον στη χρηματοδότηση του 2011 και θα μπορούσαμε ενδεχομένω και να την υπερβούμε, να δούμε με ποιο τρόπο. Βεβαίως θέλουμε να βοηθήσουμε τις κοινέ επιχειρήσεις, ε, τις διαμεθοριακές, ε, τα διαμεθοριακά εγχειρήματα, και δεν καταλαβαίνω γιατί περικόπτεται κατά 50% η συγχρηματοδότηση μελετών επιπλέον. Να τονίσουμε τι συνέβη με το ΕΦΣΥ, το οποίο δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε. Βεβαίως, συμφωνούμε ότι έπρεπε να υπάρξει μεικτή χρηματοδότηση αλλά οι μεταφορές που έγιναν για τις πιστώσεις των μεταφορών δεν ήταν οι ελάχιστες που θέλαμε. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ότι τελικά θα χρηματοδοτηθούν επαρκώς οι τομείς που μας ενδιαφέρουν. Μεταφορές και άλλοι. Και αυτά που γίνονται και για την πολιτική συνοχής. δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο γεγονό ότι μπλέκονται οι εθνικοί φάκελοι. Το θέμα είναι πώς θα συνεργαστούμε. Δηλαδή πρέπει να μην ξεχάσουμε την γραμμή ε, θαραγοθα Τερουέλ, Σαγούντο, η οποία ήταν στο ΣΕΦ 1 και χάθηκε ε, στο ΣΕΦ 2. Θα υποβάλουμε μια τροπολογία σε σχέση με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να το λόγο στην κυρία Κάπουλα Νάτρη. Κομπούλα Νάτρη, συγγνώμη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά από την Επιτροπή Ήτρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και τους τρεις εισηγητές. Εγώ εργάζομαι στην Ήτρε, οπότε θα εστιαστώ στην ενέργεια και στο ψηφιακό τομέα. Το σχέδιο έκθεση αποτελεί εξαιρετική βάση για τις συζητήσεις και για την γρήγορη ε, πρόοδο που αναμένεται και από τις δύο επιτροπές. Ε, ε, κάποια κάποια σχόλια. Ο ενεργειακός πυλώνας στον κανονισμό είναι κρίσιμη σημασία για την απαλλαγή των ενεργειακών μας συστημάτων από ανθρακούχες εκπομπές. Θα πρέπει λοιπόν να εστιαστούμε στο μέλλον, στα νέα συστήματα και όχι στα παλιά, για την επίτευξη των στόχων του Παρισιού που θα ανανεωθούν επίσης κατά τέλη του έτους ε, η κατάλληλη ώρα είναι αυτή τη στιγμή που θα πρέπει να προσέχουμε όταν βάζουμε νέους κανόνες στο ΣΕΦ. Θα πρέπει όλες οι δράσεις ε, που συμβάλλουν, να συμβάλλουν στην απαλλαγή μας από τις ανθρακούχες εκπομπές. Θα πρέπει να εστιαστούμε στα, ηλεκτρικά δίκτυα και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χρηματοδότηση για τα διασυνοριακά έργα είναι ευπρόσδεκτη, αλλά θα πρέπει να ε, γίνει σωστή χρηματοδότηση. Μπορεί να χρειαστεί περισσότερη χρηματοδότηση από αυτή που αναφέρεται στην πρόταση της Κομισιόν. Στον ψηφιακό πυλώνα θέλω να επισημάνω ότι πρόσφατα υιοθετήσαμε στην Ήτρε και στο Κοινοβούλιο ένα φιλόδοξο νομοθετικό πλαίσιο για την ε, δημιουργία ε, και την ε, επέκταση δικτύων υψηλή χωρητικότητα και των σχετικών συνδέσεων. Ε, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τώρα τη διασύνδεση και την υποδομή επενδύοντας το 5G. Πρέπει να επενδύσουμε σε κόμβους, σε δρόμους και στα βασικά δίκτυα αλλά υπάρχουν και άλλα κονδύλια για την ψηφιοποίηση όπως το Digital Europe, το EFSI και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή, να είμαστε πολύ σαφείς ε, όσον αφορά τους κανόνες, να δείξουμε ότι δεν αναμειγνύουμε διάφορους κανόνες, να δείξουμε κάποια συνοχή. Όσον αφορά τις συνέργειες, είναι κάτι στο οποίο πρέπει να συνεργαστούν οι δύο επιτροπές ε, και θα Μπορούν να προσθεθούν κάποια δευτερεύοντα κόστη χωρί προγραμματισμό, αλλά θα πρέπει να γίνουν προσεκτικά. Ευχαριστούμε κύριε Σλοτόσκη. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Να πάρω το λόγο εξ ονόματο του κυρίου Τσίλερ, ο οποίο ε, είναι ο σκιώδη συζητητή μα. Καταρχά, ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να προβληθεί σήμερα στη σημερινή συνεδρίαση. Τα βασικά στοιχεία τα οποία έχει να τονίσει είναι τα εξή. Καταρχά, ότι η ομάδα του ECR καλωσορίζει την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να μεταφερθεί το Ταμείο Συνοχή στο CEF. Ε. Είναι πραγματικά μεγάλη σημασία να συνεχίσει η ανάθεση συγκεκριμένων μέσων από το Ταμείο Συνοχή στο επόμενο πολιτέ πλαίσιο σε προγράμματα ε, μεταφορών τη CEF και σε θέματα που έχουν να κάνουν με το Ταμείο Συνοχή. 85% θα πρέπει να τηρείται ένα ποσοστό για τα δυσυνοριακά ζητήματα. Θα πρέπει πραγματικά το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο να επιτάσσεται τους ίδιους ε, κανόνες. Από πλευρά του Ταμείου Συνοχής ε, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο στη μελλοντική περίοδο όπως το προηγούμενο στο δημοσιονομικο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και αυτό το ποσό θα πρέπει να επαρκέσει σε κάθε περίπτωση προκειμένου να ολοκληρωθούν τα προηγούμενα προγράμματα υποδομών τα οποία χρηματοδοτούνται από το τρέχον Ταμείο συνοχή, Για παράδειγμα το πρόγραμμα για το Rail Baltica. Προκειμένου να υπάρχει λοιπόν καλύτερη παροχή κινήτρων και εναυσμάτων προς τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τη μεταφορά 30% του Ταμείου συνοχή, σε όλες τις χώρες συνοχή, θα γίνει εξ αρχής, από την αρχή του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου, όχι το 2024. Αυτή η πρόταση του 30% λοιπόν θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο φιλόδοξη, να έχει φτάσει και το 50% της χρηματοδότησης. μέσω διαγωνισμών. Υποστηρίζουμε λοιπόν από την ομάδα μας ε, την πρότασή σας. Ναι, παρακαλώ να ολοκληρώνετε σιγά σιγά, λέει η πρόεδρο. Αλλά το επίπεδο υποστήριξη ε, θα μπορούσε να ωφεληθεί από μεγαλύτερο ποσό στο χρηματοδότηση, 60-65%. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Τσέσακα έχει το λόγο. E, dziękuję również posłom sprawozdawcom za ich pracę nad tym raportem. Ευχαριστώ, πολύ τους εισηγητές. Χαίρομαι που οι εισηγητές επιχειρούν να απλουστεύσουν το πρόγραμμα. Το ανέφερε ο κύριος Τελίτσκα. Καθώς και τους εφαρμοστικούς κανόνες για να ενθαρρυνθεί η συνεργασία και για να μπορέσουν ε, να εργαστούν από κοινού οι τρεις ε, πυλώνες αυτού του μέσου καθώς και με άλλα μέσα όπως το Ταμείο Συνοχής. Όλα αυτά είναι θετικά. Βεβαίως, πρέπει να στηρίξουμε την κινητικότητα, την καινοτομία στον ενεργειακό τομέα και στον τομέα των μεταφορών. Όλα αυτά πρέπει να συνεργάζονται. Λοιπόν, να αναφερθώ σε ορισμένα επιμέρους θέματα. Τα επιλέξιμα προγράμματα πρέπει να ε, διευρύνουμε τα κριτήρια για αυτά τα επιλέξιμα προγράμματα για να εγκρίνουμε και κάποια διαμεθοριακά κοινού συμφέροντος. Το αναφέρει ο κανονισμός. Πρέπει να ευνοηθούν ε, τέτοια προγράμματα. Ιδιαίτερα τα διαμεθοριακά προγράμματα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αγορά της ενέργειας. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να εστιάσει επ' αυτών. Επίσης, το υδρογόνο και το φυσικό αέριο είναι σημαντικές εναλλακτικέ για το μέλλον. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι ορισμένα κράτη-μέλη όπως είπε και η κυρία Συγήτρια, σε ορισμένα λοιπόν κράτη-μέλη πρέπει να βελτιωθεί κατά πολύ η υποδομή ή απλώς δεν υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη. Κάτι άλλο που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Έχουμε και τους στόχους ε, για την κλιματική αλλαγή. Το φυσικό αέριο παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλά κράτη-μέλη, ιδιαίτερα της Ανατολικής Ευρώπης. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα της μόλυνσης. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, ή πρόεδρος. Πέτερσεν, παρακαλώ. Α, δεν είναι παρόν. Ούτε η κυρία Βιώ είναι παρούσα. Ο κύριος Θηλουάγα. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας, κύριε Θηλουάγα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να μην κρυβόμαστε. Υπάρχουν ε, πολιτικές ε, κατά της ε, διατήρησης του κλίματος και δεν πρέπει να τις κρύβουμε. Θα ξέρατε ότι πολύ πρόσφατα παρατήθηκε ο Νικολά Ιουλό που ήταν ο Γάλλος Υπουργός της Ενεργειακής Μετάβασης και τόνισε παρετούμενος ότι εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι για τις κλιματικές ανισορροπίες τα ξέρετε όλα αυτά. Αλλά όταν τα λέει κάποιο που εδώ και πάνω από ένα χρόνο ήταν υπεύθυνο για την ενεργειακή πολιτική στη Γαλλία, νομίζω ότι είναι μια ομολογία αποτυχία. Άρα θα πρέπει να αντιδράσουμε και να το δούμε το θέμα αυτό, να σκεφτούμε τι κάνουμε. Η φιλοσοφία του νέου μηχανισμού συνδέοντας την Ευρώπη είναι ίδια. Αυτό δεν βοηθάει. Και οι διακηρύξει και τα ωραία λόγια δεν πρέπει να το κρύβουν. Λένε ότι το 60% του προπολογισμού για του κλιματικού στόχου, λέγεται ότι θα είναι για κλιματικού στόχου, αλλά τι θα γίνει με το υπόλοιπο 40%. Και πώ θα καθορίσουμε εάν τα προγράμματα είναι συμβατά με του κλιματικού στόχου. Γιατί είναι πολύ ασαφή τα κριτήρια. Δεν υπάρχει σαφή ορισμό, για παράδειγμα, για το τι είναι ανανεώσιμη ενέργεια. Αυτό είναι θεμελιώδε. Ακόμη χειρότερο. Αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα γιατί, για, για το τι ακριβώς θα ε, συμπεριλαμβάνει το ανανεώσιμος. Πάνω από 5 δις ε, του υπάρχοντος ΣΕΦ που δαπανήθηκαν για ενεργειακά προγράμματα δεν δαπανήθηκαν σωστά και δεν βλέπουν να αλλάζει η προσέγγιση στο νέο πρόγραμμα. Ξεχνάμε δηλαδή τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Επίτροπος σε μια προηγούμενη ζήτηση εδώ μέσα για αυτό το μηχανισμό. Λυπούμαστε λοιπόν που το σχέδιο έκθεσης δεν διορθώνει αυτές τις ανεπάρκειες. Πρέπει να βελτιωθούν. Και μας ανησυχεί αυτή η διπλή χρήση των υποδομών, πολιτική και στρατιωτική. Θα κάνουμε τροπολογίες για όλα αυτά. Και ελπίζω να μην μιλάμε απλώς για το κλίμα, να κάνουμε και κάτι για να το προστατεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στον κύριο Κράμερ για δύο λεπτά. σα ευχαριστώ πολύ. Όταν χρειάζονται οι άλλοι τομές ε, χρήματα και πάντα από τους ε, μεταφορές. Όταν ε, ήθελε ο Γιούγκερ να χρηματοδοτήσει τα προγράμματα του, πού πήρε τα χρήματα από τις μεταφορές. Ε, και τώρα χρειάζονται τα στρατιωτικά χρήματα από τις μεταφορές. Πάλι θέλουμε να τα πάρουμε και ξέρουμε ότι και τα στρατιωτικά δεν πηγαίνουν εξαιρετικά στα κρατη και θα πρέπει να διδαχθούμε από τα σφάλματα του παρελθόντο. Να επενδύουμε μόνο αν υπάρχει συνεργασία. Δεν υπάρχει όμω συνεργασία. Ένα παράδειγμα να σα δώσω. Με ευρωπαϊκού πόρου χρηματοδοτήθηκε ο συνδρομικό διάδρομο από το Κρακοβία, Μπράσλαου, Κατοβίτσε. Έχουν ε, βελτιωθεί τα πράγματα. Οι Γερμανοί όμω ε, βγάλαν του λογαριασμού. Έχουμε ένα κενό 190 χιλιόμετρων και δεν έχει νόημα. Για το και τόσα χρόνια λοιπόν υπάρχει αυτό το κενό. Γιατί υπάρχει αυτό το μικρό κενό λοιπόν και δεν αξιοποιούμε όλο το δίκτυο. Παράλογο, αλλά αληθινό. Και το ίδιο συμβαίνει και στην Τσεχία και ε, στις Βρυξέλλες, Ανασχένα, μιλάμε για κενά 800 μέτρων μόνο για 800 μέτρα κάνουμε μία ώρα παραπάνω για να μεταβούμε από τις Βρυξέλλες τα υπόλοιπα μέρα. Δεν υπάρχει λοιπόν συνεργασία μεταξύ τα κρατών Όλα αυτά τα χρήματα λοιπόν πάνε χαμένα και το ξέρουμε από το παρελθόν τι γίνεται. Σε μεγάλα προγράμματα τα χρήματα δεν παίζουν ε, ρόλο. Κατά είναι δηλαδή η γραμμή για το Τωρίνο θα, θα έχει κοστίσει τα διπλά χρήματα, το τούνελ του Γκόταρντ, ε, το χρηματοδότησε μόνο τη Ελβετία, αλλά οι αποστάσεις αυτές ε, από τη Γερμανία και από τις άλλες χώρες δεν είναι αυτές που θα έπρεπε. Παρά το γεγονός που ξέρουμε ότι από το Μόναχο μέχρι το Μπερναμπάτης, για παράδειγμα, δεν υπάρχει ούτε μία ενιαία γραμμή Όλα αυτά λοιπόν δεν παίζουν κανένα ρόλο, γιατί το θέμα δεν είναι οι μεταφορές, το θέμα είναι τα λόμπι των τραπεζών, τα λόμπι των μεταφορών, αυτά θα πρέπει να αλλάξουν. Ε, και πριν αλλάξουν τα πράγματα αυτά, δεν θα αλλάξει και το αποτέλεσμα, γιατί οι μεταφορέ είναι ο μοναδικό τομέα ε, όπου έχουν αυξηθεί από τη δεκαετία του 90 οι εκπομπέ. Κατά πολύ τη με μεγάλα ποσοστά. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να επικεντρωθούμε και επιτέλους να υπολογίσουμε και το κόστος των συνεπειών σε ό,τι αφορά το κλίμα, το περιβάλλον. Να ξέρουμε όμως τι, όσο πιο λίγα κάνουμε σήμερα, τόσο πιο πολύ θα κληθούμε να πληρώσουμε αύριο. Και εδώ, στον τομέα των μεταφορών, μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος και την προστασία του περιβάλλοντος. Και παράλληλα αυτά, λείπει συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει κατεπηγόντως. Και φυσικά επενδύουμε μόνο σε νέα προγράμματα. Δεν επενδύουμε στη συντήρηση των παλιών ε, προγραμμάτων. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι στο Βέλγιο υπάρχει, υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Φυσικά γίνεται εξοικονόμηση πόρων, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στις υποδομές, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ότι λείπουν τα καινούργια project, καινούργια έργα. Το πρόβλημα είναι η συντήρηση των παλιών έργων. Και θα πρέπει, θεωρώ, να διδαχθούμε πιο πολύ από τα σφαλμάτα του παρελθόντο. πριν αρχίσουμε και σπαταλάμε δισεκατομμύρια εδώ και εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Μαρσελέζη, καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μα και έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ του εισηγητές και ιδιαίτερα την κυρία Φιρκούνεν, την εισηγήτρια τη ΣΥΤΡΕ. Συμφωνώ με πολλέ προτάσει. που περιλαμβάνουν η πρόταση, ιδιαίτερα για τη διαφάνεια, για το κόστος την αύξηση των ε, συνεργασιών, της κοινή δράσης, για να επιτύχουμε την ψηφιοποίηση. Νομίζω ότι η πρόταση της Επιτροπής έχει επίσης σωστές προτάσεις. Μια ειδική πρόταση για το κόστος που έχουν να κάνουν με το κλίμα. Αυτό πρέπει να βοηθήσει να εκπληρώσουμε τους στόχους των ε, Παρισίων και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο νομοθετικό τμήμα του κειμένου. Πρέπει τα λόγια να γίνουν πράξη και πρέπει να έχουμε και σαφή κριτήρια που να επιτρέπουν το δημόσιο χρήμα που θα χρησιμοποιηθεί στο ΣΕΦ τις επόμενες δεκαετίες να χρησιμοποιηθεί με υπεύθυνο τρόπο. Δεν θέλουμε ε, νέα προγράμματα για ε, ορυκτά καύσιμα. Δεν θέλουμε και άλλους ε, πετρελαγωγούς. Πρέπει να προωθήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα. Και επίσης θέλουμε να προωθήσουμε τα διαμεθεωριακά προγράμματα ανανεωσίμων. Ε, πρέπει λοιπόν να περάσουμε πολύ περισσότερο στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μικρού επίπεδου, περίπλοκα αλλά καινοτόμα. Πρέπει να γίνουν αναγκαίες μελέτες για να έχουμε και τις αναγκαίες ιδιωτικές επενδύσεις και τα joint venture. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε το ίδιο και τα ΕΦΗ δίκτυα να αναφερθεί σαφώς στην έκθεσή μας τη Ήτρε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συνεργασία με τους εισηγητές γιατί πιστεύω ότι είναι όντως το κείμενο αυτό επαρκές για να κάνουμε τα λόγια πράξη ούτως ώστε επιτέλους, επιτέλους όπως είπαμε και χθε, να περάσουμε σε υψηλότερη ταχύτητα για να αξιοποιήσουμε σωστά τους πόρους μας για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ κύριε Μαρκελέση. Η κυρία Νταμάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους συναδέλφους. Οι υποδομές ε, ε, των μεταφορών στην Ευρώπη ε, θα πρέπει να εστιαστούν στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ασφάλεια των πολιτών μας. Επιτρέψτε μου συνάδελφοι να πω ότι για μας ε, ακόμα είναι ανοιχτή η πληγή μετά από την κατάρρευση της γέφυρας ε, στη Γένοβα με 43 θύματα. Συμφωνώ με όλους σας ε, και πιστεύετε κι εσείς, είμαι βέβαιη, ότι δεν είναι δυνατόν να πεθαίνει κόσμος από κατάρρευση γεφυρών ε, και ελλείψεις υποδομών στην Ευρώπη. Η ασφάλεια λοιπόν πρέπει να είναι βασικός παράγοντας στη νέα πρόταση του ΣΕΦ και οι απαιτήσει ασφαλείας θα πρέπει να είναι πρωταρχικοί παράγοντες για την αξιολόγηση των προγραμμάτων νέων ή υπάρχουσων υποδομών. Ωστόσο, ο προπολογισμό που προτείνει η Κομισιόν φαίνεται να απέχει πολύ από τα απαραίτητα οικονομικά κονδύλια για την ολοκλήρωση μέχρι το 2030 του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Τα ποσά που διατίθενται σε όλα τα κράτη-μέλη για τις μεταφορές ε, είναι μόλις 12,8 δισεκατομμύρια σε σχέση με το 30,6 που απαιτείται και για τη στρατιωτική ε, κινητικότητα και τη συνοχή. Η Ιταλία συμβάλλει σημαντικά στον προπολογισμό της Ένωσης. Ωστόσο, στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο ε, χρηματοδότησε στο Νότο με δικά της κονδύλια ε, πολλές υποδομές. Θέλουμε μες τα επόμενα χρόνια λοιπόν μια πιο ίση κατανομή. Αν προσθέσουμε σε αυτό ότι οι επενδύσεις μπλοκάρουν από δημοσιονομικές ε, δεσμεύσεις που περιορίζουν τις ε, δυνατότητες δαπάνης, εμείς θα απαιτήσουμε μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές οι επενδύσει αυτέ. Επίση, ζητάμε μεγαλύτερη καθαρότητα όσον αφορά τα ποσοστά συγχρηματοδότηση και δράσεις σωστές. Θα κάνουμε και κάποιες αλλαγές στον έλεγχο ε, των ε, ε, χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο για τις χρηματοδοτήσεις και να υπάρξουν και κατεξουσιοδότηση πράξεις για το στρατιωτικό σκέλος. Ευχαριστούμε κυρία Ανταμάτο. Δίνω το λόγο στον κύριο Τέλουσκα που εκπροσωπεί τον κύριο Πέτρεσεν. Κύριε Πρόεδρε, το συγγνώμη που δεν μπορεί να παραβρεθεί εδώ ο συνάδελφο και που τον έδρασα πιο νωρί. Δυστυχώ, λοιπόν, ο συνάδελφο δεν μπορεί να παραβρεθεί εδώ σήμερα. Και λυπάται ιδιαιτέρω. Γιατί το ΣΕΦ θεωρεί ότι αποτελεί μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη. Μια ευκαιρία για να απαντήσουμε στις δεσμεύσει ε, της Συμφωνία του Παρισιού σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος. Επίση, εκτιμά την εργασία των εισηγητών για το σκέλος της ενέργειας του ΣΕΦ θα ήθελε να καλωσορίσει και τις τροπολογίες και έχει να τονίσει τρία στοιχεία. Καταρχάς, τροπολογία 2 σε ό,τι αφορά τις υποδομές αερίου για τις πιστεύει έντονα ότι θα πρέπει να είναι υψηλό το επίπεδο της ε, φιλοδοξίας για την τροπολογία 23, για τα διασυνοριακά προγράμματα και έργα. Πιστεύει ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τη φιλοδοξία πάνω από το 10% και για την συγχρηματοδότηση για την τροπολογία 43 τονίζει ότι χρειάζεται ε, δέσμευση του δημοσίου τομέα προκειμένου να υπάρξουν και ιδιωτικέ επενδύσεις. Αυτά και ζητά και πάλι συγγνώμη που δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα στη συνεδρίαση. να δώσω το λόγο και πάλι στην κυρία Νταμάτο που εκπροσωπεί τον κύριο Ταμπουράνο, ο οποίος δεν μπορεί να παρευρεθεί για το θέμα της ενεργείας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο για τον συνάδελφο Ντάριο Ταμπουράνο που είναι συνεισηγητής ε, στην Επιτροπή Ήτρε και ζητά συγγνώμη που απουσιάζει αλλά ήθελε να συμβάλλει. Ευχαριστεί τους συζητητές για το σχέδιο έκθεση όπου βρίσκει με μεγάλη το ευχαριστή κάποιες βελτιώσεις σε σχέση με την πρόταση τη Κομισιόν όπως η αναφορά στην ενεργειακή απόδοση και ε, την κυβερνοασφάλεια ω στόχοι που πρέπει να επιδιωχθούν στον τομέα της ενέργειας και ε, των ψηφιακών. Αναφέρεται και βελτίωση των δικτών παρακολουθησής και ελέγχου των επενδύσεων του προγράμματος. Θέλει να ενισχυθούν αυτές οι βελτιώσεις, ιδίως όσον αφορά το κλιματικό και περιβαλλοντικό κομμάτι ώστε να εφαρμοστούν ε, τα λόγια και οι υποσχέσεις που δόθηκαν στο Παρίσι ε, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους που μόλις εγκρίθηκαν στη Δεσμή για την Ενέργεια, αποφεύγοντας ε, την θανάσιμη παγίδα της επιστροφής στις ορεκτές πηγές ενέργειας. Θέλουμε λοιπόν να προτείνουμε πρώτον αύξηση του ποσοστού του προϋπολογισμού για τους κλιματικούς στόχους από 25% στο 30-40%. Δεύτερον, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του ΣΕΦ για τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το κλίμα, ε, καθιστώντας τις δεσμευτικές αν είναι δυνατόν και αποκλείοντας τις προτάσεις που αντιτίθεται αυτή τη αρχή. Επίση, ε, να μειωθούν οι επενδύσεις για τα ορεκτά ε, καύσιμα, να φτάσουμε στο 0 μέχρι το 2050 να ακολουθήσουμε το καλό παράδειγμα λοιπόν των ταμείων συνοχής, του Ταμείου Συνοχής να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση με την αρχή Energy Efficiency First στο πλαίσιο της ε, ενεργειακής διακυβέρνησης και συμπεριλαμβάνοντας και προγράμματα ενεργειακής απόδοσης που χρηματοδοτούνται μέχρι του ΣΕΦ, να διευκολυνθούν οι επενδύσεις στις υποδομές όπως τα Smart Grid, να βελτιωθεί η κλιματική ο κλιματικός έλεγχος των προγραμμάτων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν απαλήφοντα το greenwashing ε, που σχετίζεται με τις ορυκτέ πηγές και βελτιώνοντα του δείκτε παρακολούθηση των προγραμμάτων υποδομών που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα. Ο συναδέλφο, θα υποβάλει σχετικέ τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Νταμάτο, δίνω το λόγο στον συναδελφό μου τώρα για να διαχειριστεί ε, τη συζήτηση. Ε, Έχετε τον λόγο κύριε Ρούμπεκ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε Ντελή. Επειδή η Ήτρε ε, συμμετέχει στη διοργάνωση αυτής της συνεδρίασης, είναι σημαντικό τώρα να ακούσουμε και τους ευρυπλέον ομιλητές. Επειδή ενεγράφησαν πάρα πολύ, είμαι υποχρεωμένος ε, να δώσω στον καθένα ένα λεπτό για να τελειώσουμε στις 12.30. Ο πρώτος ο κύριος Ρικέ. Ένα λεπτό. Άρα ένα μόνο θέμα. Χρειαζόμαστε πάρα πολλές υποδομές. Και τα κράτη-μέλη ούτε τις συντηρούν, ούτε αναπτύσσουν ε, το ΣΕΦ έχει επιτύχει και δεν είναι επαρκή η χρηματοδότησή του. Έγιναν πολύ παραπάνω προτάσεις για χρηματοδοτήσεις από αυτό. Έχουμε λοιπόν τεράστιες ανάγκες ακόμη. Είναι περιορισμένος φυσικά ο προπολογισμό. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο να αυξηθεί ο προπολογισμό. Και το γεγονός ότι αξιοποίησαμε 10 δις από την ε, πολιτική συνοχή ε, για το συνδέοντα στην Ευρώπη, όπως αναγνώρισαν και τα κράτη-μέλη, λειτουργήσε σωστά. Γι' αυτό θα προτείνω σε μια άλλη τροπολογία 20 δις από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας να, περάσει, να περάσουν, όπως ακριβώς κάναμε για το Ταμείο Συνοχής, στο συνδέοντα στην Ευρώπη. Έτσι πιστεύω ότι θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους μας. Ευχαριστώ πολύ. Κέλλη. Σον Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές. Το ΣΕΦ είναι πολύ επιτυχημένο και θα συνεχίσει πιστεύω να είναι και το στηρίζω πλήρως. Ο Πάβελ είπε ότι πρέπει να χρηματοδοτήσουμε και τις συνδρομικές ε, μεταφορές γιατί ορισμένες ε, είναι ζημιογόνες. Πολλά έχει κάνει το ΣΕΦ για τους σειροδρόμους και δεν νομίζω ότι έχει έννοια να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε ζημιογόνες επιχειρήσεις. Αν υπάρχουν ε, κοινωνικοί λόγοι για να γίνεται κάτι τέτοιο, να το κάνουν τα κράτη-μέλη, όχι η Ένωση. Δεν έχουμε επαρκεί πόρου. Για να κάνουμε αυτά που χρειάζεται, χρειάζεται να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, και να αναπτυχθούν τα PCI. Νομίζω ότι η ε, ο, οι αύξησης των μεταφορών, ιδιαίτερα των οδικών μεταφορών, δεν είναι πλέον βιώσιμη. Πρέπει να ε, φύγουν οχήματα από τους δρόμους. Δεν έχουμε κάνει επαρκή. Πιστεύω ότι μόνο έτσι θα επιτύχουμε τους κλιματικούς στόχους. Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς πόροι. Πρέπει να προωθήσουμε τα έργα κοινού ενδιαφέροντο. Αυτά είναι τα θέματα για μας. Ευχαριστώ πολύ. Γκάλα. Ευχαριστώ πολύ. Στο υπάρχον πρόγραμμα έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο μέτρο. 20%, 20 επιδότηση για την αντιμετώπιση του, των θορύβων, ιδιαίτερα για να ε, εισαχθούν ορισμένα είδη φρένων που κάνουν λιγότερο θόρυβο. Όμως ο στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί, λέει η Κομισιόν. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει αυτή η επιδότηση και στο μέλλον. Αυτό στηρίζω. Κάτι άλλο. Η στρατιωτική κινητικότητα. Χαίρομαι πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το περιέλαβε στο κείμενο. Ξέρω ότι οι συγκητές κάπως το αποδυνάμωσαν, αλλά εν πάση περιπτώσει εντάξει, μας ικανοποιεί. Ξέρουμε ότι είναι η διπλή χρήση, βασικά πολιτική και στρατιωτική όταν χρειάζεται. Στην άλλη, Κράμερ. Πρέπει να ενισχύσουμε τη στρατιωτική κινητικότητα. Έτσι θα μπορέσουμε να κλείσουμε τα... τις τρύπες αυτές, για παράδειγμα, μεταξύ Κότμπους και Σιλεσίας. Νομίζω ότι αν βάλουμε το Wilhelmshaven ή το Rotterdam ή την Αμβέρσα ε, στους τομείς αυτής της στρατιωτικής κινητικότητας θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Γιατί η πραγματικότητα είναι Φανβρεμία. Ευχαριστώ κυρία Φαν Μπρέμπτ. Ευχαριστώ. Να τονίσω ένα σημαντικό θέμα. Ενεργειακό θέμα. Οι περισσότεροι παρόντες νομίζω θα μπορουσαμε να βοηθησουμε γιατι η πραγματικοτητα ειναι οπως ειναι η κυρια φανμπρεμπτ ευχαριστω να τονισω ενα σημαντικο θεμα ενεργειακο θεμα οι περισσοτεροι παροντες νομιζω θα συμφωνουσαν ότι δεν είναι πολύ αποτελεσματικό να επιδοτούμε και στο μέλλον μέσω δημοσίου χρήματος τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Όλοι μιλήσαμε για την κλιματική αλλαγή. Το κάνουμε στο παρελθόν. Υπενθυμίζω ότι 60% του ΣΕΦ ενέργεια πήγε στο φυσικό αέριο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Και υπήρχαν ε, βάσιμοι λόγοι γι' αυτό. Πρέπει να αυξήσουμε την ε, ανεξαρτησία μας από τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να περάσουμε από μια μεταβατική περίοδο. Αλλά είμαι τελείως πεπισμένη ότι τελείωσε αυτή η περίοδος. Και ξέρετε ότι η Συμφωνία των Παρισιών είναι το πλαίσιο για το ΣΕΦ ενέργειας. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριό μας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Ευχαριστώ, κύριε ε, Ριβ... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και θα ήθελα καταρχάς να επισημάνω ότι υποστηρίζω τις ε, ε τροπολογίες που θέλουν να περιορίσουν στο 10% τη χρηματοδότηση. Οι επιδοτήσει θα πρέπει να παραμένουν θέμα κεντρικό σε ό,τι αφορά τις μεταφορές ε, που χρειάζεται μακροπρόθεσμες επενδύσεις και μεγάλη συμμετοχή του δημοσίου κλάδου σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι θέλουμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα, θέλουμε να κοιτάξουμε λοιπόν τη συμμετοχή των κρατών μελών και πώς καταφέτουν προτάσεις που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Χαίρομαι λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη και τοπικές και περιφερειακές διαστάσεις σε ό,τι αφορά την ε, πρώτερη έγκριση από πλευρά των κυβερνήσεων. Αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει και τα, με τα δίκτυα αυτά. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες και τις ενέργειες που θα υποστηριχθούν, είναι απαραίτητο να προσθέσουμε και τις δράσεις που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα της ποιότητας των ε, υπηρεσιών για να υπάρξει καλύτερη σύνδεση μεταξύ των περιφερειών και των αστικών κέντρων και της υπέτρου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Φαντεκάμπο, επόμενος. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ να ευχαριστήσω τους τρεις εισηγητές. Προσπαθούμε να συμπληρώσουμε τη χρηματοδότηση της, τρίτης δεκαετίας. Αυτό είναι πολύ απαραίτητο και κρίσιμο. Τέσσερις παρατηρήσεις. Καταρχάς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε σε εφορία, γιατί τα δίκτυα αυτά πάνε πίσω. Όλοι μιλούν για την ενεργειακή καμπή, για το model shift, αλλά ο σιδηρόδρομος και η ιστορική ναυσιπλοεία μειώνονται. Ελπίζω λοιπόν το ΕΛΚΑ να καταθέσει τις σωστές τραπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Δεύτερο σχόλιο, η συμμετοχή του Ταμείου Συνοχής. Καταλαβαίνω ότι θέλει εξυγχρονισμό και πιο πολύ ανταγωνισμό και νέε προδιαγραφέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά φροντίσουμε η συμμετοχή από το Ταμείο Συνοχή να μην διακυβεύεται και να μην υπονομεύεται, γιατί εκεί βλέπω κάποια στοιχεία που με ανησυχούν. Όσο πιο πολύ περιορίζουμε το Ταμείο Συνοχή και τη συμμετοχή του, τόσο πιο δύσκολα θα τα πράγματα. Συμφωνώ με τον Γκάλερ και τον Ταλίτσκα που λένε ότι ε, στρατιωτική πόρη και διπλή χρήση. Ωραία. Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως, Πρόεδρε, είναι το εξής, ότι η στοχοθεσία στον κανονισμό ε, ΣΕΦ είναι πολύ ασαφέ. Αυτό τι θα σημαίνει, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει μικρότερο λόγο και όλο πιο πολλά κενά θα γεμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα επόμενα 7 χρόνια. Το θέλουμε αυτό. Και τέλος θα καταθέσουμε μια τροπολογία για το πότε θα γίνουν οι διαγωνισμοί. Αυτό κάθε φορά παραμένει ασαφές και για κάποια έργα πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για τους διαγωνισμούς. Πρέπει να ξέρουμε πότε και πώς θα προετοιμαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντεμόντα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συζητητές ε, και για αυτό το κείμενο που μας έχουν παρουσιάσει. Θέλω να υπογραμμίσω πόσο σημαντικός είναι ε, για τον τομέα των μεταφορών ε, η υλοποίηση των δικτύων TNT. Για ολόκληρο το δίκτυο. Είναι λοιπόν σημαντικό να δώσουμε προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των έργων υποδομών των διασυνοριακών, ε, όπως για παράδειγμα μεταξύ Τωρίνου και Λιών. Εκεί θα πρέπει να δείξουμε κάποια συνοχή. Δεν μπορούμε να λέμε από τη μια ότι θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές και από την άλλη να μην δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργηθούν τα κομμάτια που θα βοηθήσουν στην καλύτερη βιωσιμότητα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Και τώρα για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Γένοβα που υπενθυμίσατε κυρία Πρόεδρε στην αρχή της συνεδρίασης πρέπει οπωσδήποτε να, δώσουμε, να καθορίσουμε κάποιες προτεραιότητες. Καλή είναι η συνδεσιμότητα βέβαια αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να έρχεται η ασφάλεια των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και γιατί τηρήσατε και το χρονικό όριο. Ο κύριος Βαντάλ είναι ο επόμενος. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Τρία σημεία έχω να κάνω. Καταρχά χρηματοδότηση, προπολογισμό θα βγει ένα μεγάλο κράτο μέλο το 2019 να μην αυξηθεί ο προπολογισμό. Δεύτερον, στρατιωτική χρήση, διπλή χρήση. Όποιο γνωρίζει την αεροπορία ξέρει ότι δεν λειτουργούν τα θέματα διπλή χρήση και ότι είναι αναποτελεσματικά τα αεροδρόμια αυτά. Ας μην ξεκινήσουμε λοιπόν να προσθέτουμε τέτοιες θετικές χρήσεις για την παλιά δόξα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα βιώσιμοι τομείς όπως ε, οι σιδηρόδρομοι και άλλοι τομείς να ε, προθεθούν. Και εδώ ανησυχώ ιδιαίτερα γιατί πολύ φοβάμαι ότι τα προγράμματα ιστορικής ναυσιπλοείας όπως το Φρίσλαντ για παράδειγμα θα αναβαγίσουν γιατί θα δοθεί πιο πολύ προσοχή στις οδικές μεταφορές οι οποίες λοιπόν δεν μπορούν να τα από μόνες τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ ο εισηγητής από τις ΑΦΕΤ και ο, της ΕΝΤΕ, ο κύριος Καστάλτο. Δύο λεπτά έχετε στη διάθεσή σας, κύριε Καστάλτο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Μηχανισμός Σύνδεσης της Ευρώπης, το ΣΕΦ, χρηματοδοτεί προγράμματα που έχουν στόχο τη σύνδεση της Ευρώπης ευρυζωνικά στις μεταφορές και στην ενέργεια. Σε αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να ξεχνάμε τους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Τομείς ε, που ε, συζητώνται όλο και περισσότερο και σε εμά και που σημειώνουν τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Ω εισηγητή ε, στη ΣΕΝΤΕ για το στρατιωτικό σκέλο, ε, θέλω να σα πω προ τα που κινούνται οι δικέ μου τροπολογίε. Πρώτα απ' όλα, σε τι επικεντρώνεται η στρατιωτική κινητικότητα. Δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς στενή συνεργασία με το μη στρατιωτικό σκέλος. Με άλλα λόγια, οικονομικά δεν θα είχε νόημα να δημιουργούνται υποδομές αποκλειστικά στρατιωτικής χρήσης. Πιο σωστό, χρηστό οικονομικά, είναι να βρούμε τις μη στρατιωτικές άξονες, σε ε, λιμάνια, αεροδρόμια, που μπορούν να εξυπηρετήσουν και στρατιωτικά μέσα, δηλαδή διπλής χρήσης. Να... Χρειάζεται λοιπόν στενή συνέργεια με τον πολιτικό τομέα και με την υποστήριξη των διαφόρων τοπικών κοινωνιών με έργα συμμετοχικά και συνεργατικά χωρίς αποκλεισμούς. Πιστεύω ότι η διπλή χρήση και οι σχετικές υποδομές πρέπει να θεωρούνται σημαντικές. Αναφέρομαι τώρα στα work criteria του άρθρου 13, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα στρατιωτικά πρότυπα μπορούν να προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια των εν λόγω υποδομών. Τέλος, η στρατιωτική κινητικότητα πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή και να έχει, δίνει ιδιαίτερη προσοχή και στο περιβαλλοντικό σκέλος, να τηρεί όλα τα απαραίτητα πρότυπα σε σχέση με την ρήπανση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. Το δεύτερο κομμάτι είναι η πολιτική συγκυρία στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Η κρίση που ε, ταλανίζει την Ευρώπη απαιτεί ε, να δείξουμε όραμα, να αποφύγουμε περαιτέρω ε, προβλήματα επιχειρησιακά, δηλαδή να εντείνουμε τις στρατιωτικές μας δυνατότητες ε, για όλους τους σκοπούς και για φυσικές καταστροφές. Δηλαδή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις πιθανές μελλοντικέ απειλές. Το στρατιωτικό σκέλος, λοιπόν, γεωγραφικά θα πρέπει να είναι ισορροπημένες, να επιτρέπεται η κίνηση προσωπικού και μέσων ε, στον βόρειο νότιο άξονα και στον άξονα Δύσης Ανατολής. Ευχαριστούμε. Από την Επιτροπή των Περιφερειών η Ιζαμπέλ Μποδονέ. είναι η συγγήτρια και έχει επίσης δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτά τα δύο πολύτιμα λεπτά που προσφέρετε στην Επιτροπή των Περιφερειών. Πράγματι οι περιφέρειές μας, οι πόλεις μας είναι, παίζουν σημαντικό ρόλο ε, για την αλλαγή των μεταφορών προς μια καθαρή κινητικότητα και συμφωνώ με την κυρία Ρεβονταλόν η οποία μίλησε για το ρόλο μας ως περιφερειών και κοινοτήτων. Παρακολουθούμε στενά τις προτάσεις σας. Έχουμε αλλάξει το πρόγραμμα εργασιών μας για να συντονιστούμε με εσά. Είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο, πιστεύουμε, και η Επιτροπή των Περιφερειών να συνεργαστούν ώστε να ε, αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες των πολιτών εκεί όπου έχουμε εκλεγεί. Ω εισηγήτρια, ε, με επιταχυμένη διαδικασία, σήμερα το απόγευμα θα προεδρεύσω μια συνεδρίαση των ενδιαφερομένων και την εκθεσή μου θα την υποβάλω σήμερα. Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου μπορώ να συμπεριλάβω εκεί τροπολογίες για τη βελτίωση της έκθεσης και δικές μου και τέλος η έκθεση αυτή θα υποβληθεί στην Ολομήλεια της Επιτροπής των Περιφερειών 8 και 9 Οκτωβρίου. Πριν κλείσω, θα ήθελα να πω ότι όπως είπε ο κύριος Ντομινίκ Ρικέ, ε, είναι πολύ καλό αυτό το εργαλείο ε, για μας. Ναι, θα είναι χρηστή η διαχείριση του δημοσίου χρήματος, αλλά δεν έχουμε επαρκή φιλοδοξία εδώ. Η Ευρώπη θα βελτίωνε την αξιοπιστία της ε, αν επένδυε περισσότερο για μεταφορά των εμπορευμάτων από τα εκατομμύρια φορτηγά ε, που μολύνουν τους δρόμους μας στους σιδηροδρόμους. Ας κάνουμε προτάσεις λοιπόν μαζί για να ολοκληρώσουμε αυτούς τους διαδρόμους, να τους βελτιώσουμε και ώστε πράγματι να ε, μεταβούμε στις σιδηροδρομικές μεταφορές ε, κάτι που θα επηρεάσει θετικά το κλίμα και θα μας βοηθήσει να τηρήσουμε και τις συμφωνίες του Παρίσιου όπως είπαν πολύ προαλήσαντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η DG Move θα εκφραστεί. Ο κύριος Όλιβερ Ζέλερ. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ε, τρεις συνσηγητές για την εργασία τους και για τη στήριξη σε μεγάλο βαθμό που δίνουν στο ΣΕΦ. Νομίζω ότι οι γενικές γραμμές ε, του σχεδίου έκθεσης βρίσκουν σύμφωνη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τα σημεία ακριβώς όπου λέγεται ότι πρέπει να ενισχυθεί ή να βελτιωθεί το κείμενο. Πρώτα απ' όλα κοινέ προσπάθειες. Πρέπει να έχουμε όλες τις ε, δυνατότητες ανοιχτές. Δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα και κοινών προγραμμάτων εργασίας για ορισμένα θέματα. Ο συνδυασμός είναι περίπλοκο θέμα, το blending. Δεν μην ξεχνάμε βεβαίως ότι αυτό το blending θα υποκαταστήσει τις επιδοτήσεις το μεγαλύτερο τμήμα του προπολογισμού του ΣΕΦ θα πάει σε παραδοσιακές επιδοτήσεις. Αλλά οι δύο τελευταίες προσπάθειες συνδυασμού που κάναμε στις δύο τελευταίες προκηρύξεις στις μεταφορές μας έδωσαν ε, την εμπειρία ότι βοηθάει για να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια διατύπωση που να είναι συμβατή με τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό. Έχουμε λοιπόν κάποια τεχνικά θέματα για αυτό το θέμα του συνδυασμού που πρέπει να δούμε. Η συγχρηματοδότηση των μελετών. Μπορεί να φαίνεται μικρή σημασία, αλλά δεν είναι. Μέχρι στιγμή 50% και για τους τρει τομεί μπορεί να αποτελέσει ποσοστό συγχρηματοδότηση. Πιστεύω ότι έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε ε, τη σωστή χρηματοδότηση των μελετών. Και δεν είναι θεωρητικές μελέτες. Είναι μελέτες ε, περιβαλλοντικής επίπτωσης, είναι μηχανολογικές μελέτες. Πρέπει λοιπόν να διατηρηθεί το 50% του ποσοστού χρηματοδότησης στους ε, βιομηχανικούς τομείς. Οι προτεραιότητες των μεταφορών. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ της συντήρησης και, της, ε, του εξυγχρονισμού του δικτύου. Πάρτε ένα άλλο μικρόφωνο. Λοιπόν, άλλο μικρόφωνο. Προτεραιότητα στον τομέα των μεταφορών. Πρέπει να υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ εξυγχρονισμού και ανάπτυξης του δικτύου. Πολλά υπόθηκαν για το κλίμα. Είδατε την πρότασή μας. Δεν νομίζουμε ότι η συμπερίληψη των αεροδρομίων ε, ε, είναι, ε, βοηθάει την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Συμφωνούμε με το Κοινοβούλιο να βάλουμε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες ε, στο μέσο για την στρατιωτική κινητικότητα και να υπάρχουν περισσότερες εγγυήσεις ότι οι επενδύσεις ε, διπλής χρήσης μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Πρέπει λοιπόν να διατηρηθεί η αναλογικότητα. Δεν ε, θα πρέπει όλα τα τμήματα του TNT να μπορούν να συμπεριληφθούν στα θέματα στρατιωτικής κινητικότητας. Πρέπει να δούμε τι είναι θέμα κινητικότητας και τι είναι θέμα υποδομών. Τέλος, για την ψηφιοποίηση. Υπόθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει ακριβέστερη διατύπωση των ε, προγραμμάτων κοινού συμφέροντος στον τομέα αυτό. Αλλά δεν θέλουμε διατύπωση να περιορίσει το εύρος ε, των προγραμμάτων που θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε. Βεβαίως είμαστε ανοιχτοί για μια αναδιατύπωση και με χαρά να το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την έκθεσή σας και προσβλέπουμε στην περαιτέρω συνεργασία με τους εισηγητές στις επόμενες φάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό για τον κάθε εισηγητή. Παρακαλώ. Ο κύριος Μαρινέσκου. Δεν έχει σχόλια. Πολύ καλά. Κύριο Τελίτσκα. Δύο λεπτά δηλαδή έχω εγώ. Όχι, όχι. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο να κάνω. Καταρχά. Καταρχά το ερώτημα των διαφορετικών ε, λειτουργιών και των τρόπων. Σε ό,τι αφορά τη πλωτέ οδού. Θα πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα αυτό. Αυτό να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς ε, σχετίζεται η συνεργασία μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Ξέρω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα αν υπήρχε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων για να προετοιμάσουν ε, την ε, φάση τη εφαρμογή σε ό,τι αφορά την εποπτεία από πλευρά του Κοινοβουλίου. Το ανέφερε και ο Βιμ και άλλοι ενδεχομένω. Σίγουρα θα το παρακολουθήσουμε αυτό και θα το φροντίσουμε αυτό για την επόμενη περίοδο, αλλά προσπαθούμε ήδη να ενισχύσουμε την εποπτεία. Για τι ε, μελέτε, αντέδρασε η Επιτροπή. Αυτό είναι ένα τρόπο να τα κοιτάξουμε τα πράγματα. Το άλλο θέμα είναι το εξή. Αν θέλω να εφαρμοστεί ένα πολύ σημαντικό ε, έργο, ως ε, κράτος μέλος στη φάση αυτή όπου δεν είναι ακόμα τόσο μεγάλη η πόρη θα μπορούσε να προβώ ως κράτος μέλος σε επενδύσεις. Το θέμα λοιπόν είναι να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Και τέλος σε ό,τι αφορά το στρατητικό σκέλες, αυτό που είπε και ο κ. Κράμερ αλλά και άλλοι, για τις αναποτελεσματικότητες που υπάρχουν. Δεν παίρνουμε τον προπολογισμό από τις μεταφορές. Δεν αφαιρούμε από τις μεταφορές Αντιθέτως, έχουμε επιπλέον προπολογισμό, επιπλέον πόρους. Θέλουμε απλά να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα πάνε σε αυστηρός και αμυγός στρατιωτικούς στόχους, ότι υπάρχει διπλή χρήση. Και δεν μιλάμε την ενίσχυση, για την ενίσχυση, για παράδειγμα, της άμυνας, της παρουσίας μας, της κάπου. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε στην Νότια μια κατάσταση και να πρέπει να μεταφέρουμε ε, βαρύ εξοπλισμό στο σημείο αυτό. Α, υπό το πρίσμα αυτό θα σας παρακαλούσα να το κοιτάξετε αυτό και αξίζει τον κόπο και πιστεύω ότι ε, θα μας βοηθήσει. Ευχαριστώ και συγγνώμη που μίλησα παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βερικονένα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Και φυσικά είναι πολύ ελπιδοφόρα αυτή η συζήτηση, γιατί φαίνεται ότι όλοι συμφωνούν για την σημασία του προγράμματος ΣΕΦ και όλοι προφανώς θέλουν τα χρήματα αυτά να δαπανηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό προφανώς και είναι ελπιδοφόρο για το μέλλον μας και προσβλέπουμε στις ε, τροπολογίες σας και στις μελλοντικέ παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει η κυρία Τελή, θα ήθελα να ευχαριστήσω πριν τη λήξη της συνεδρίασης τους τρεις συζητητές για την εργασία την οποία κάνουν. 13 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. 9 Οκτωβρίου είναι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας και παρακαλώ να με ακούσετε μέχρι τέλους. Τα συμπεράσματα τα μας ε, τρομάζουν, αλλά μπορεί να έχουν και ένα ψήγμα ελπίδα. Σήμερα λοιπόν καταλάβαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε όλοι και ζούμε πάνω σε ένα ηφαίστειο σε ό,τι αφορά το κλίμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να βγάλουμε την ουρά μας απ' έξω. Θα πρέπει να έχουμε ένα συνολικό όραμα μεταξύ της ενέργειας, των μεταφορών, το ψηφιακό σκέλος δεν μπορούμε να βάλουμε σε κουτάκια το όραμά μας. Θα πρέπει να φροντίσουμε ότι οι επενδύσεις να μην γίνονται διπλά. Δεν υπογράψαμε τη συμφωνία της COP21 για να κάνουμε πίσω στις επενδύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί εισηγητές. Είσαστε πραγματικά σε επαγρύπνηση και πέρυσι τη συνεδρία